Αγαπητοί συνάδελφοι, τα πρακτικά της συνεδρίας αυτής θα εγκριθούν στην επόμενη συνεδρία του Κοινοβουλίου και τα ψηφίσματα αυτά θα διαβιβαστούν στους ε, αποδέκτες τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και εύχομαι σε όλους τους βουλευτές και τους υπαλλήλους μια καλή επιστροφή. Α, ο κύριος Όντι για διαδικαστικό θέμα προηγουμένως.